στην αρχή, οι ελληνικές αρχές μου υπέβαλαν δύο αιτήματα άρσης ασυλία των κυρίων Σωτηρίου Ζαριανοπούλου και Γεωργίου Γραμματικάκη στα πλαίσια ε, ποινικών διαδικασιών. Το αίτημα, σύμφωνα με τον κανονισμό, θα αποσταλεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η ομάδα των Σοσιαλιστών